και τον συγχαίρω γι' αυτό, το Κοινοβούλιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τους Ευρωβουλευτές διαπιστώνει ότι η έδρα του κ. Κατρούγκελου είναι κενή από τις 27 Ιανουαρίου και το ανακοινώνει αυτό στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.